Ε, της Γαλλικής Δημοκρατίας μου έστειλαν δύο αιτήματα άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας ε, για την κυρία Μαρίν Λεπέν και για την κυρία Μαρή Κριστίν Μπουτονέ στο πλαίσιο δικαστικών ερευνών που ξεκίνησαν από το οικονομικό τμήμα του Δικαστηρίου των Παρισίων ε, σύμφωνα με τον κανονισμό. Αυτά τα αιτήματα θα σταλούν στην Νομική Επιτροπή του